υποφέρουν από τις συνέπειες αυτής της απαράδεκτης σύγκρουσης. Ευχαριστώ κύριε Ποτότσνικ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Επτά όπως είπα είναι την προτάση ψηφίσματος για τις οποίες θα κάνουμε ψηφοφορία μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων. Το επόμενο θέμα είναι η κλιμάκωση της βίας στο Μεξικό. Και θα ακούσουμε τους συντάκτες των ψηφισμάτων με πρώτο τον κύριο Γιουρικού Ατόντο. Για ένα λεπτό. Για τρία λεπτά. Sí. Señor Presidente. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι το Μεξικό είναι μια μεγάλη δημοκρατία, μια δημοκρατία που εξελίχθηκε προεδευτικά την τελευταία 20 Είναι μια χώρα φίλη, φίλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα με την οποία έχουμε συνάψει συμφωνία στρατηγικής σύνδεσης. Επίσης το Μεξικό δίνει μια σκληρότατη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Σήμερα όμως εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλούμε για το Μεξικό στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο κεφάλαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί διαπιστώσαμε μια σημαντική έξαρση της βίας, μια κλιμάκωση της βίας ε, με θύμα το μεξικανικό λαό. Και υπάρχουν επανειλημμένες και σοβαρότατες καταγγελίες για καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μεξικό. Το ψήφισμα που υπέβαλαν οι μεγαλύτερε ομάδε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα εγκρίνουμε σήμερα στηρίζεται στο σεβασμό, στηρίζεται στη συνένεση και αναγνωρίζει αυτό το πλαίσιο που σας περιέγραψα και παροτρύνει το Μεξικό να συνεχίσει τις προσπάθειές του να συνεχίσει την διαμόρφωση ενός κράτους δικαίου και μιας τέλειας δημοκρατίας. Ζητά όμως από το Μεξικό και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Πρώτον, να εξασφαλίσει την άσκηση ε, της ε, ελευθεροτυπίας, γιατί έχουν διαπιστωθεί επιθέσεις ε, εναντίον δημοσιογράφων να εξασφαλίσει την προστασία των ενώσεων και σωματείων που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί υπάρχουν απειλέ και επιθέσει κατά οργανώσεων που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να εξασφαλίσει τα θύματα τη βία, που είναι κυρίω γυναίκε, γιατί υπάρχουν και γυναικοκτονίε, και να παταχθεί η ετοιμορρησία. να επανέλθει η ασφάλεια στη χώρα του Μεξικού. Αυτό ζητούμε ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το, Ευρωπαϊκό. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο θα πάρει τώρα η κυρία Ρενάτε Βέμπερ για δύο μισή λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, τη βδομάδα αυτή γιορτάσαμε την Διεθνή ημέρα της γυναίκας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, αναρτήσαμε αφήσει σε όλες τις γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης λέγοντας «Ναι, μπορεί να σταματήσει η βία κατά των γυναικών». Σήμερα μιλούμε για τη βία στο Μεξικό και είναι λογικό να θυμηθούμε ότι οι γυναίκες του Μεξικού, αυτόχθονες ή όχι, είναι τα θύματα που τη χάνουν τις λιγότερες προστασίες από τις τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές του Μεξικού. Οι γυναίκες του Μεξικού είναι θύματα πάσης μορφής βίας, της οικογενειακής βίας, της σεξουαλικής βίας, βασανιστήριων, είτε από στρατιωτικούς είτε από αστυνομικού, μέχρι και θύματα γυναικοκτονίας. Μέχρι σήμερα η απάντηση των μεξικανικών αρχών ήταν αποτελεσματική. Γι' αυτό και ουσιαστικά μιλούμε για παντελή ατιμορρησία των ενόχων. Το ψήφισμά μας ζητά από τη μεξικανική κυβέρνηση να καταπολεμήσει τις γυναικοκτονίες. Είναι βάναυση αυτή η ορολογία, αλλά είναι σωστή, γιατί σχεδόν όλες οι δολοφονίες κατά των γυναικών ε, μένουν ατιμόρυτε. Για παράδειγμα, στην πολιτεία του Μεξικού τα τελευταία τέσσερα χρόνια καταδικάστηκαν μόνο 11% των ε, εγκληματιών που δολοφόνησαν ε, εκατοντάδες γυναίκες. Ταυτόχρονα φαίνεται ότι οι γυναίκες είναι τα θύματα που προτιμάει και το δικαστικό σύστημα. Πώς εξηγείτε ότι δύο αυτόχθονες γυναίκες, η Αλβέρτα Κάνταρα και η Τερέσα Κοσάλες, καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 21 ετών και μέχρι στιγμής έχουν περάσει πάνω από τρία χρόνια στις φυλακές επειδή σε, μία, ε, σε ένα σούπερ μάρκετ έκλεψαν φρούτα. Μακάρι ο δικαστής που θα αποφασίσει, θα απειληθεί σε μία εβδομάδα την προσφυγή, το ένδικο μέσο, την έφεση, να αντιληφθεί την γελιότητα της κατάστασης και την αδικία της ποινής. Ελπίζω ότι οι Μεξικανοί νομοθέτες πολύ σύντομα θα βελτιώσουν το γενικό νόμο πρόσβαση των γυναικών σε μια ζωή χωρίς βία, θα στοιχειοθετήσουν τις ε, μορφές βίας και θα προβλέψουν τους μηχανισμούς για να εφαρμοστούν αυτές οι νομοθετικέ διατάξεις. Επίσης, η οικογενειακή βία και ο, βιο, ο, ο βιασμός και με στο γάμο είναι ποινικά κολάσιμες πράξεις καταγγέλουμε και απορρίπτουμε τη βία κατά των γυναικών. Και αυτό το θέμα θα πρέπει να γίνει στοιχείο διαπαιδαγώγησης και να συμπεριληφθεί ήδη από τα πρώτα χρόνια της σχολικής εκπαίδευσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπίλαν, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Οι αρχές του Μεξικού και κυρίως ο πρόεδρος Φελίπε Καλτερών ε, έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια ολόκληρα αιμοσταγή αγώνα κατά των λαθρεμπόρων ναρκωτικών με θύματα πολλούς στρατιώτες και με λίγες νίκες. Για παράδειγμα έχουν συλληφθεί κάποιοι επικεφαλής καρτέλ και ε, πολλά εκτάρια μαριχουάνας και οποίου έχουν παροπλιστεί ενώ έχουν φυλακιστεί πολλοί όσοι συμμετείχαν σε, τέτοιες, σε, καλλιέργεια ή διάθεση ναρκωτικών. Βέβαια το εμπόριο ναρκωτικών αποφέρει τεράστια κέρδη. Δυστυχώς η κυβέρνηση του Μεξικού δεν έχει καταφέρει να εκριζώσει το εμποριο ναρκωτικων αποφερει τεραστια κερδη Δυστυχώ η κυβερνηση του ναρκωτικών. Και η διαφθορά επίσης είναι τεράστια, ακόμη και δικαστών αστυνομικών, γι' αυτό και συνεχίζεται ο, ο Μόνο το Οκτώβριο πέρυσι είχαμε πάνω από 6.000 θύματα και πολύ συχνά ε, χάνουν τη ζωή τους και ε, δημοσιογράφοι. 13 μονοδολοφονίες είχαμε το 2009. Χρειάζεται λοιπόν μια παγκόσμια υποστήριξη για να κερδίσει το Μεξικό αυτό το σκληρό αγώνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπιέλα. Ε, ο κύριος Φίσσα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, στο Μεξικό υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα ναρκωτικών και ελευθερμπορείων ναρκωτικών που δημιουργεί και παράγει βία. Ο πρόεδρο Καλτερών προσπάθησε με πυγμή και στεναρά να εκριζώσει αυτό το φαινόμενο και τη μάστιγα, χρησιμοποιώντα και τι ένοπλε δυνάμει με πολύ σημαντικά ε, αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την καταστροφή ναρκωτικών, την κατάσχεση όπλων και την ε, σύλληψη ενόχων. Επίσης έγιναν δεκτές ε, όλες οι στάσεις της ε, Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ακόμη και σε ό,τι αφορά την ανάκριση και τις έρευνες που γίνονται για τη δράση του στρατού. Επίσης η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης ε, σε θέματα ασφάλειας και δικαιοσύνης και ξεκίνησε μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος προκειμένου να αποκατασταθεί η διαφάνεια και να τιμωρούνται οι αυτούργοι των εγκλημάτων με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δείξουμε την αλληλεγγύη μας προς το Μεξικό στον αγώνα του κατά των ναρκωτικών και να υποστηρίξουμε τον πρόεδρο Καλντερών στην επιθυμία του να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα. Επίση, θέλω να εκφράσω την ε, ικανοποίησή μου για, την, για το ψήφισμα αυτό που προσυπογράφουν οι μεγαλύτερε ομάδε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Η κυρία Βερσία για να Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι παραβιάσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα χειροτερεύουν συνεχώς στο Μεξικό σύμφωνα με, τα, με τις ΜΚΟ. 800 δολοφονίες αποδόθηκαν στα καρτέ των ναρκωτικών ε, για το 2009 στην περιοχή κυρίως της Τσιχουάουα. Ο Καλτερόν έχει στείλει χιλιάδες στρατιώτες σε όλη τη χώρα, αλλά οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευράς των στρατιωτικών δυνάμεων και των δυνάμεων καταστολής αυξάνονται. Οι ΜΚΟ μιλάνε πλέον για εγκλήματα από πλευράς των κρατικών δυνάμεων, εις βάρος ιδιαίτερα των γυναικών ηθαγενών ημί. Συναντήθηκα με κάποιες από αυτές τις γυναίκες στο Σαν Σαλβαντόρ Αντένκο που βιάστηκαν και βασανίστηκαν από τις δυνάμεις καταστολής. Αυτοί οι οποίοι διέπραξαν τις πράξεις αυτές το 2006 παραμένουν ατιμόρυτοι. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να συμφωνήσουμε με αυτά που λέγουν οι μεξικανικές αρχές, των οποίων, οποίας μάλλον, των οποίων οι υπάλληλοι παραβιάζουν συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ κύριε Βερσιά. Για 1,5 λεπτό η κυρία Λοχπίλερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι εικόνες των αιματηρών ε, συγκρούσεων στους δρόμους ε, του Μεξικού ε, για τα ναρκωτικά ή φόνη βάρος γυναικών, συνήθως εργατριών στη βόρεια χώρα με τον τίτλο «Γενοκτονία» έχουν συγκλονίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και, μας, ε, και έχουν ε, περιληφθεί μέσα σε μία έκθεση. Πλην όμω και παρά τι συνεχιζόμενε ε, παραβιάσει των δικαιωμάτων, φαίνεται ότι η μεξικανική κυβέρνηση δεν είναι σε θέση ή δεν έχει τη βούληση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κατάσταση. Ούτε, η, ούτε επαρκεί η καταπολέμηση των συμμοριών των ναρκωτικών. Η παρουσία της αστυνομίας παντού, οι αρμοδιότητες των στρατοδικείων, η ατιμορρησία για τα εγκλήματα που έχει διαπράξει οποιοδήποτε όργανο της τάξης ή των όπλων δυνάμεων οδηγούν σε μια συνεχή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχιζόμενα εγκλήματα από το στρατό. Η κυβέρνηση παραγνωρίζει τη σημασία ακόμη πολλών ε, εγκλημάτων όπως σε παραδείγματι ε, βλέπουμε με την προσπάθεια από την κυβέρνηση εχθές ακόμη ε, ανακοινώθηκε από τον Υπουργό από έναν Υπουργό του Μεξικού ότι θα καταβάλουν σημαντικά χρηματικά ποσά στα θύματα των παθόντων μόνο και μόνο για να τους πλήσουν το στόμα απαιτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να καθυστερήσει την υπογραφή της συμφωνίας με το Μεξικό όσο συνεχίζονται ...η παραβιάση των αυτοπινών δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Λόχ Πίλερ. Τώρα συνεχίζουμε με τις ομάδες. Παρέμβαση εκ μέρους της ομάδας του ο κύριος Πρέντα. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η κλιμάκωση της βίας στα στις περιοχές του Μεξικού που βρίσκονται κοντά στη, στα σύνορα με τι ΗΠΑ και ιδιαίτερα στην, πόλη Σουηδά Χουάρε έχει οξυνθεί ιδιαίτερα, είναι ανησυχητική. Βλέπουμε αύξηση των εγκλημάτων που σχετίζονται με τον θεμποριό των ναρκωτικών και τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών τον συνοδεύει και ένας ακύρωτο πόλεμος μεταξύ των συμμοριών των ναρκωτικών με πολλά θύματα. βλέπουμε στην περίπτωση του Μεξικού ότι απαιτείται να καταβληθούν προσπάθειες να αναλάβουμε δράση αποφασιστικά έτσι ώστε να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτά τα δεινά. Πρέπει να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα στη μεξικανική κυβέρνηση, να την πιέσουμε, να εκριζώσει την εγκληματικότητα και να ε, βοηθήσει τον λαό της. Πρέπει να ενθαρρύνουμε και τις μεξικανικές αρχές επίσης να εδραιώσουν το κράτο δικαίου, να προχωρήσουν ρύθμιση του συστήματο τη δικαιοσύνη και τη αστυνομία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκόμε, για ένα λεπτό. Η βία στο Μεξικό συνδέεται με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών αλλά και τι κοινωνικέ ανισότητε που επιδεινώνονται από την οικονομική κρίση. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί η ετοιμορρησία, να επενδύσουμε στο δικαστικό σύστημα και να φέρουμε ενώπιον των δικαστηρίων του ενόχου. Πολλές νέες γυναίκες εργαζόμενος έγιναν θύματα της βίας των λαθρεμπόρων ναρκωτικών. Η Σιουδάδ Χουάρε είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα των γυναικοκτονιών. Επίσης, ε, η φαλοκρατική νοοτροπία αφήνει ατιμόρυτους ε, τους αυτουργού και φέρνει στο βωμό το, της αδικίας πολλά θύματα και δημοσιογράφους. Θέλουμε να υποστηρίξουμε το Μεξικό για να ε, υποστηρίξει τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί αυτοί είναι ε, οι άνθρωποι που δίνουν μάχη υπέρ της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, γιατί χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα δεν νοείται ούτε κράτος δικαίου ούτε δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο κύριος Τσαρνέτσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πριν από λίγο άκουσα στην αίθουσα αυτή μια έκκληση να μην υπογραφεί η Συμφωνία σύνδεση με το Μεξικό. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί πριν από λίγο είπαμε ότι επενούμε και το, είπε, και, ε, το είπε και πολλοί προλαλήσαντε. Επικροτούμε την προσπάθεια του πρόεδρου του Μεξικού ε, να καταπολεμήσει τις μαφίες και τους λαθρεμπόρους των ναρκωτικών. Θα πρέπει να επικροτήσουμε, να επιδοκιμάσουμε τις προσπάθειες της μεξικανικής κυβέρνησης Φυσικά θα πρέπει με τα ξερά να κάνουμε και τα χλωρά, να ρίξουμε το, νερό, το παιδί με τα, βρώμικα νερά και να δούμε, να καταλάβουμε την κατάσταση μιας χώρας που εδώ και δεκαετίες ε, έχει να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο κύμα ε, οργανωμένου εγκλήματος ε, από τις μαφίες. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον πρόεδρο και την κυβέρνηση του Μεξικού σε αυτόν τον αγώνα κατά του οργανωμένο εγκλήματο. Βέβαια, θύματα αυτού του αγώνα πολλέ φορέ είναι και οι δημοσιογράφοι. Θα πρέπει να τονίσουμε τη δική του συμμετοχή. Σίγουρα δεν θα πρέπει να γίνεται διακριτική μεταχείριση βάρο των δημοσιογράφων. Ευχαριστώ. Ο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ακόμη και σήμερα το πρωί το Ευρωπαϊκό Συνδικάτο Ελεκτρολόγων περικυκλώθηκε από αστυνομική δύναμη 100 με 200 αστυνομικών. Το συνδικάτο αυτό ανήγγειλε για τις 16 του μηνός ε, γενική απεργία και ο κύριος Ντομίνγκο Αγιλάρ Βάσκας, ο πρόεδρος αυτού του συνδικάτου, συνελήφθη. Είναι πραγματικά συνταρακτική αυτή η κατάφορη παραβίαση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων εκ μέρους των μεξικανικών αρχών. Μιλούμε για την ατιμορρησία ε, στη μεξικανική κυβέρνηση, με ατιμορρησία των ε, στρατιωτικών, των αστυνομικών και ε, διαπιστώσαμε μια αναποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των ναρκωτικών. Γιατί η κυβέρνηση του Μεξικού επιτίθεται ταυτόχρονα κατά των λαθρεμπόρων ναρκωτικών, αλλά επιτίθεται και κατά των συνδικαλιστών. Η Μεξικανική Δημοκρατία δυστυχώς ολισθαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Φυσικά θα πρέπει να καταγγείλουμε τέτοιες παρεκτροπές και να ζητήσουμε από τη μεξικανική κυβέρνηση να γίνει πιο αποτελεσματική και να δείξει περισσότερη πυγμή απέναντι στους λαθρεμπόρους αρκωτικών και να είναι πιο ελαστική απέναντι στα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Ευχαριστώ. Εξαντλήσαμε του ομιλητέ εκ μέρου των ομάδων. Τώρα η κυρία Κόρχολα, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω τη σημασία του ψηφίσματό μα για δύο κυρίω λόγου. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με, τις, με τα καρτέλ των ναρκωτικών στο Μεξικό, τα, στα οποία οφείλεται ο θάνατος 15 συνολικά χιλιάδων ανθρώπων Ιδιαίτερα στι περιοχές κοντά στα σύνορα με τι ΗΠΑ, όπου δεν μπορεί ούτε ο στρατός ούτε η αστυνομία να ελέγξουν την κατάσταση. Η ευθύνη λοιπόν για την ε, ε, συνεχιζόμενη αυτή αταξία, για τα προβλήματα αυτά τα συνεχιζόμενα, ανήκει πραγματικά στα καρτέλ. Επίσης η Εθνή Αμνηστία έχει ε, καταδικάσει την ατιμορρησία σε σχέση με τις επιθέσεις από πλευράς οργάνων της ε, τάξης ε, του Μεξικανικού κράτους εις βάρος αγωνιστών των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας κατά της ατιμορρησίας. Και εν ώψη και της ε, Συνόδου Κορυφής μεταξύ Πολιτειών και Μεξικού ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Τιτσάου για ένα λεπτό. Η κυβέρνηση του Μεξικού θα πρέπει να αναλάβει και να φέρει πέρα τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει σε σχέση με το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στις πόλεις της Τιχουάνα και της Σουδάδ Χουάρες είναι από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον κόσμο το 2009 με εκατοντάδες νεκρούς. Ε, τι εκατοντάδες, χιλιάδες νεκροί στα πλαίσια της, ε, της δραστηριότητας των συμμοριών ναρκωτικών. Οι γυναίκες και οι νέοι φυσικά φύγονται πρώτοι από τη βία και την κατανάλωση των ναρκωτικών. Η οικονομική κρίση βέβαια στο Μεξικό θα οδηγήσει και σε κοινωνικές συγκρούσεις και είναι αυτό που οδηγεί στην κατανάλωση των ναρκωτικών. 7,5 εκατομμύρια νέοι ζουν στο Μεξικό εκτός του επίσημου συστήματος παιδείας. Δεν υπάρχει διάλογος ανάμεσα στους νέους και στην κυβέρνηση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση και η κατάσταση στον τομέα της ασφαλείας. Ευχαριστώ τον κύριο Τσιτσάου. κύριος τώρα για ένα λεπτό. Πρόεδρε. Συχνά εδώ συζητούμε προβλήματα από τις δικτατορίες ανά τον κόσμο, αλλά το Μεξικό δεν είναι δικτατορία, είναι δημοκρατία. Έχουμε να κάνουμε μονομενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά αυτό δεν στιγματίζει το Μεξικό ως χώρα. Στιγματίζουμε εδώ τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει μια μεγάλη δημοκρατία εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και δεκαετίες. Ένα μας στο οποίο πρέπει να δώσουμε λύσεις και θεραπείες κατάλληλες. Ο πρόεδρος Καρτερών είναι αυτός ο γιατρός ο οποίος θα δώσει τις θεραπείες και τα φάρμακα. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να παίξουμε το δικό του ρόλο, πρέπει να παίξουμε το ρόλο του ιατρού, αλλά να στηρίξουμε το γιατρό με ένα ενισχυμένο δημοσιονομικό μέσο, με ενισχυμένη παρουσία δική μας, με στήριξη του κράτους δικαίου, των κρατικών δομών, με την υποστήριξη που θα προσφέρουμε στο Μεξικό για να ανοικοδομήσει το κράτος του και να αποφύγει την αποδιάρθρωσή του και με τη στήριξη που θα προσφέρουμε για την καταπολέμηση των συμμοριών των αρκομτικών. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πόσλτ και τώρα περνάμε στη δικασία Catch the Eye. Βίλαν Μόντ, παρακαλώ. Όλοι ανησυχούμε με την κλιμάκωση της βίας στο Μεξικό και στις Χιδαδ Πάντως ε, εγώ έχω εμπιστοσύνη στι μεξικανικέ αρχέ και στα μέτρα που υιοθέτησαν και που θα αντιμετωπίσουν αυτή την περίπλοκη κατάσταση. Επίση, υποστηρίζω τη στεναρή μάχη που δίνει ο πρόεδρο Καλτερών κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, μια παγκόσμια μάστιγα που μα επηρεάζει όλου. Όλοι θα πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτό το σκληρό αγώνα και να υποστηρίξουμε του μεξικανικού θεσμού. Τα τελευταία δέκα χρόνια το Μεξικό βάδισε το δόμο τη δημοκρατία και τη ε, χρηστή διακυβέρνηση και το Μεξικό ανέλαβε περισσότερες ευθύνες και σε παγκόσμιο επίπεδο και συμμετέχει ενεργά στις επιχειρήσεις ε, του G10 και των Ηνωμένων Εθνών. Εγώ είμαι υπέρ της ε, στρατηγική σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση με το Μεξικό, που τελικά το πετύχαμε το 2008. Ελπίζω στη διάσκεψη κορυφή τη Μαδρίτης να θετηθεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα κοινή δράση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά να κάνει με το Μεξικό και σε διμερέ επίπεδο, αλλά και σε πολυμερέ επίπεδο, για να αντιμετωπίσουμε από κοινού προκλήσει και απειλέ συμπεριλαμβανομένων του λαθρεμπόριου ναρκωτικών και άλλων μορφών οργανωμένου εγκλήματο. Ευχαριστώ τον κύριο Μιλάν Μον και έτσι. ο κύριο Τάνακ παρακαλώ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για πολύ μακρύ διάστημα ήταν το Μεξικό ο κύριος αγωγός διέλευσης των ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Και έτσι οι σχέσεις του... Το Μεξικό το ίδιο έχει εδρεωμένα μέσα, δρομένες μέσα στην ε, επικράτειά του πολλές και μεγάλες οργανώσεις λαθρεμπορίου των ναρκωτικών. Τα χρόνια έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και με την εγκληματικότητα σχετική με τα ναρκωτικά, αλλά και με τους αποτρόπαιους άλλους φόνους, των οποίων πέφτουν θύματα όχι μόνο οι νέοι οι και τα παιδιά, αλλά ιδιαίτερα, ιδιαίτερα άλλες ομάδες όπως τη δημοσιογράφη. Βλέπουμε ε, ορισμένες περιοχές του Μεξικού να έχουν βρεθεί τελείως εκτός ελέγχου. Οι αρχές δεν είναι σε θέση να συγκρατήσουν τη βία. Ο πρόεδρο Καλτερών χρειάζεται υποστήριξη, κάνει προσπάθειε για την αναδιάρθρωση του συστήματο αστυνομία, τη διαφθορά, των σχέσεων, τη διαπλοκή με τα καρτέλ των ναρκωτικών και θεωρώ ότι ήταν αιτιολογημένη η απόφασή του να χρησιμοποιήσει προσωρινά το στρατό για την αποκατάσταση της τάξης. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε τώρα η διαδικασία του Catch the Eye και θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Ποτότσινικ για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια αύξηση των εγκλημάτων χωρίς προηγούμενο έχει δημιουργήσει αισθήματα ανασφάλειας στον πληθυσμό. Ανησυχεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζουμε ότι οι μεξικανικές αρχές αντιμετωπίζουν με σοβαρό τρόπο το πρόβλημα και έχουν πάρει αρκετά μέτρα. Ο πόλεμος του Πρόεδρου Καλτερών, εναντίον του εγκλήματος του οργανωμένου είναι βασική προτεραιότητα. Πέρα από την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων, το Μεξικό κάνει τεράστιες προσπάθειες στον τομέα της προστασίας της τάξης, της ένομης τάξης. Ήδη από τον Αύγουστο του 2008 υιοθετήθηκε μία σειρά μέτρων η οποία βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των κατασταλτικών και δικαστικών δυνάμεων της χώρας. Υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν με αυτά τα μέσα τα ενδυμικά προβλήματα στον τομέα των ποινικό, αν και η πλήρης εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι μακροχρόνια. Κάνει προσπάθειες στο Μεξικό για να ανταποκριθεί επίσης και στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οργανωμένο έγκλημα, ελευθερία του τύπου, ελευθερία έκφρασης. Είναι θέματα τα οποία φέρνουν στην επιφάνεια και στην προσοχή μας οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Γι' αυτό έχει υπάρξει και μια ειδική εισαγγελία στο Μεξικό για τα εγκλήματα εις βάρος των δημοσιογράφων το 2009. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα ακόμα, αλλά υπάρχουν ε, και μέτρα και στον τομέα της εκπαίδευσης και γενικότερα γύρω από την υπόθεση αυτή. Ο νέος ομοσπονδιακός νόμος, σαν παράδειγμα για την σωματεμπορία, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Καλείται λοιπόν το Μεξικό να υιοθετήσει μια οργανωμένη πολιτική, να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και η ακαιρεότητα και προστασία αυτών που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τμήμα θα έλεγα της έκθεσης που παρουσιάζει το Μεξικό στην περιοδική συνάντηση που οργανώνουν τα Ηνωμένα Έθνη. Πρόσφατα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που έγινε σε επίπεδο κορυφής το Νοέμβριο του 2009 ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Μεξικό στις Βρυξέλλες τέθηκε το θέμα της βοήθειας και συνεργασίας και οργανώθηκε στο Κανκούν ένα διεθνές σεμινάριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την όμιμη χρήση της βίας για την προστασία των και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταλήξαμε σε ένα κοινό κείμενο για τον έλεγχο και τις ευθύνες των τοπικών δυνάμεων καταστολής. Και το κείμενο αυτό κατετέθηκε στην ε, τοπική βουλή. Έχουν επίσης υιοθετηθεί και ομοσπονδιακοί νόμοι για την μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και γενικότερα θεωρούμε ότι η νέα στρατηγική συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει. Οι στρατηγικοί εταίροι συνεχίζουν τους διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να υπάρξει ένας επίσημος διάλογος γύρω από τα θέματα της ασφαλείας όπως επίσης να υπάρξει και ενισχυμένη συνεργασία και με τη Europol, τη Eurojust και, τα... και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιμετώπισης Κατάχρησης Ναρκωτικών κτλ. Όλοι υποστηρίζουμε το σχέδιο 4 με 7 για την ενίσχυση της συνεργασίας με τις αστυνομικές αρχές του Μεξικού και μέχρι το, την επόμενη φάση 11 με 30. Είναι φανερό ότι το Μεξικό αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα ούτε ιδεώδης η κατάσταση, αλλά επίσης πρέπει να πούμε ότι το Μεξικό δείχνει τη θέληση να δημιουργήσει μια σωστή πολιτική δημόσιας ασφάλειας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Επίτροπε κύριε Πετώση. Ε, έχουν υποβληθεί τα ψηφίσματα που θα ψηφίσουμε στο τέλος της συζήτησης. Το επόμενο θέμα είναι η Νότιος Κορέα. Η θανατική ποινή κρίνεται παράνομη. Θα ήθελα καταρχήν να δώσω